Presidente. Buenas noches, colegas. Buenas noches, señor comisario. Καλησπέρα σας. Η μερίσια διάταξη προβλέπει αυτή τη στιγμή τη δήλωση Επιτροπής Εξέβρεση Λύσεων για την Άκαμψη της Οικονομίας στα κράτη, με, στα κράτη της ε, Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης, τα οποία είναι μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο λόγος των ε, Επίτροπο, ήθελα να πω, πήγα να πω αντιπρόεδρο, εν πάση περιπτώσει, στον ε, Επίτροπο κύριο Αλμούνια, μέλο Επιτροπής. Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, η οικονομική κρίση